κριτικής επί τη βάση ε, μελλοντικής αναλύσεως και ρεαλιστικών προσδοκιών. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δεχούχτ. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητέ εξορμώσει των Επιτροπών. Ο κύριο Μάρτιν από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.